ε, συναδέλφων ε, μου κοινοποίησαν πως ε, λόγω της κακοκαιρίας της προηγούμενης εβδομάδας υπλήξαν πάρα πολλοί πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είχαμε πλημμύρες, σφοδρές γενοπτώσεις και Νομίζω πως ε, όπως αυτό το ζήτησαν και οι ομάδες θα συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να εκφράσω εξ ονόματος σώματος την αλληλεγγύη μας ε, στους ε, πληγέντες και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να βοηθήσει γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία. 22 Ιανουαρίου Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την δεύτερη διάσκεψη για το μέλλον της Συρίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. όπου θα έχουμε τους εκπροσώπους ε, του Συριακού Καθεστώτος και της Συριακής Αντιπολίτευσης με τους διεθνούς εταίρους με στόχο να βρεθεί ένας τρόπος να τελειώσει ο εμφύλιος και να σχηματιστεί μια μεταβατική κυβέρνηση. Η δύσκολη κατάσταση στην ε, Συρία βεβαίως δυσκολεύει τη διεξαγωγή Τη διάσκεψης αυτή, η οποία όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από όλου του συμμετέχοντες να μην αναβάλουν την διάσκεψη, αλλά να παραβρεθούν. Τα... Οι κοινοβουλευτικέ ομάδες ενέκριναν επίση το αίτημα αυτό ομοφόνο και βέβαια θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσοχή τις εξελίξεις στην Συρία μέχρι να σταματήσει η σύγκρουση. Κυρίες και κύριοι, με πληροφόρησαν πως ο συνάδελφος Μπροκ ε, δέχθηκε επίθεση από τον, λεκτική επίθεση από τον ε, Πρωθυπουργό της ε, Ρουμανίας για κάποιες δηλώσεις του που έκανε σχετικά με την μετανάστευση εντός της Ένωσης και τον παρομοίασαν με Ναζί. Ανεξαρτήτως ε, του περιεχόμενου των δηλώσεων του κυρίου Μπρόκ, θεωρώ πως είναι απαράδεκτο πρώτο να γίνονται τέτοιες συγκρίσεις και βεβαίως δεύτερον νομίζω πως δεν τίθεται ζήτημα για την ακαιρεότητα του κυρίου Μπρόκ. Περνάω τώρα στις ανακοινώσεις. Το πρόγραμμα, το σχέδιο χρονοδιαγράμματος του 2015 είναι στην διάθεσή σας. Εγκρίθηκε η πρόταση αυτή από την διάσκεψη των Προέδρων. Τρίτη 14 Ιανουαρίου είναι προθεσμία για τροπολογίες και τετά